αλλά η μητρική μου γλώσσα είναι τα ουγγρικά. Βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα στην Ανατολική Ευρώπη, βλέπουμε ότι είναι ανησυχητική η κατάσταση και η κατάσταση όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στην Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πούτιν δεν είναι οι καλύτερες και αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί τους Σλοβάκους. Εμείς ε, θελήσαμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρήσαμε ότι θα μας προστατεύσει την δημοκρατία. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές ε, αξίες οι οποίες στήθεται σε κίνδυνο σήμερα λόγω ακριβώς της ανόδου του λαϊκισμού. Αναφέρομαι σε ανθρώπους και στη ρητορική ε, όπως ο κύριος Φάραντς και τι σκέφτεται σε σχέση με την ανεξαρτησία της Σκοτίας και το δημοψήφισμα εκεί. Σας ευχαριστώ λέει ο Λέμε ομιλίες ενός λεπτού και πρέπει να είναι ομιλίες ενός λεπτού και πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες. Ο κύριος Σάιμον έχει το λόγο τώρα. Η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει περισσότερους πόρους ε, στην μεταποίηση ή στη μηχανική. Το να κάνει κανείς ε, πράγματα ε, με τα χέρια δεν είναι τόσο της μόδας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε καλοί στην Ευρώπη, ιδίως σε σχέση με άλλες περιοχές, αλλά και στα δυτικά Midlands έχουμε πολλές τέτοιες βιομηχανίες οι οποίες εξάγουν σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει όμως ε, να είναι ε, όλο και καλύτερη στελέχωση αυτών των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δεξιότητες ε, του εργατικού δυναμικού αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η εγγύηση για την νεολαία θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρά τις πιέσεις, αυτό που χρειάζονται οι νέοι είναι ποιοτικέ, βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίμων. Κύριος Κούτσενγιουκ έχει το λόγο. Κούσνιουκ. Ο κύριος Κούσνιουκ. Δεν εμφανίστηκε ο κύριος Κούσμιουκ. Ο κύριος Σταρβάτη έχει το λόγο. Ούτε και ο κύριος Σταρβάτη είναι εδώ. Ο κύριος Γιούρεκ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι χώρες μας ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή στις ευρωεκλογές από τους Πολωνούς πολίτες την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ήρθαν τρία προεξέχοντα άτομα, ο Ρόμαν Βότσεκ και Εξέγος, που ήταν ε, προσκυνητές και ήταν πεζοί γυρίζοντας όλη την Ευρώπη. Πέρασαν από την ε, Ιρλανδία, το Μοντεκασίνο, μετά την Πολωνία και μετά ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουν την ειρήνη στον κόσμο και πάνω απ' όλα για να δουν τι γίνεται με την κατάσταση αυτών οι οποίοι θα πρέπει να ήταν τα θύματα της ε, σύραξης στην Ουκρανία. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους και ελπίζω ότι μπορούν να είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Ευχαριστώ κύριε Γιούρεκ. Ο κύριος Τσίτσι. Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι στη διάρκεια της θητείας μας δεν θα έχουμε νέους συναδέλφους εδώ, διότι διαπραγματεύσεις ε, ε, ενταξιακές που δίκησαν πάνω από πέντε χρόνια σταμάτησαν. Εγώ δεν θεωρώ όμω ότι θα έπρεπε να σταματήσει η διαδικασία τη διεύρυνση, αλλά να ενταθεί, διότι χώρε από την Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν ε, τι δικέ του φιλοδοξίε, τι δικέ του επιθυμίε και βέβαια κυρίω μιλώ για Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία. Σερβία, ε, Μαυροβούνιο, Αλβανία. Υπήρξαν ε, συζητήσεις το καλοκαίρι και με τους πρωθυπουργού των χωρών αυτών και φαίνεται ότι η κατάσταση στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο είναι τέτοια που θα ήθελαν πραγματικά να έχουν εδώ εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια γι' αυτό φυσικά και πρέπει να εκπληρώσουν όλα τα προαπαιτούμενα. Πιστεύω όμως ότι τα Βαλκάνια χρειάζονται ειρήνη και η ειρήνη είναι ουσιαστικά ταυτόσιμη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τους δώσουμε μια σαφή προοπτική λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιακοβτσίτς ο κύριος Χουαρίστη Αμπαουτσολός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, το μεγαλύτερο μέρος της βασικής κοινωνίας έχει δύο προτεραιότητες, την ειρήνη και την αυτοδιάθεση. Και μια σαφής εκλογική πλειοψηφία το έχει κατάδειξει αυτό, όπως δείχνει και η παρουσία μας σε αυτό το κοινοβούλιο είναι η στιγμή που θα πρέπει να ανακτήσουμε όλα τα δικαιώματά μας ως άτομα αλλά και ως λαός και ιδίως το δικαίωμα των Βάσκων να αποφασίσουν την τύχη τους. Η λύση στην ε, διαμάχη με τη χώρα των Βάσκων είναι και θέμα της Ευρώπης. Αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παροτρύνει και πάλι τις Γαλλικές και ισπανικέ κυβερνήσει να είναι θαραλέ, να υποστηρίξουν τις λύσεις και όχι να διατηρήσουν πολιτικές και στρατηγικές του παρελθόντο που βασίζονται στο όχι και στην αντεκδίκηση. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει πάλι στην Ισπανία στην, ε, ε μια δίκη εναντίον 28 νέων και επίσης υπήρξε ε, και βία κατά ε, συγγενών κρατουμένων. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε μαζί με την κοινωνία των Βάσκων για την αυτοδιάθεση και την ειρήνη. Και είμαστε δεσμευμένοι να το πράξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χουαρίστη. Ο κύριος Μαραγκάλ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για λίγα δευτερόλεπτα στα καταλανικά. Un ben Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, με ακούτε? Θα συνεχίσω στα ισπανικά, λέει Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε 24 παρεμβάσεις. Αν χρησιμοποιείτε μία άλλη γλώσσα, <clears throat> τότε δεν πρόκειται να σας μεταβράσουμε. Αν θέλετε λοιπόν, να, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό θα έκανα, κύριε Πρόεδρε. Η Καταλωνία είναι ένα παλαιοευρωπαϊκό έθνος, γνωρίζει τι είναι και τι θέλει να πετύχει. Η Καταλωνία έχει μια ισχυρή σαφή φωνή για μια δημοκρατική οδό για την νομιμοποίηση της απόφασης που θέλει να πάρει για το δικό της το μέλλον. Η Ευρώπη δεν ε, θα πρέπει ούτε μπορεί να μην ενδιαφερθεί για την φιλοδοξία που εκφράζουμε ελεύθερα εμείς ένας ιστορικός λαός ε, για μια κοινωνία δεσμευμένη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αλλάζει. Η Σκοτία Καταλωνία είναι θετικά παραδείγματα αυτής της βαθιάς αλλαγής, ε, μιας αλλαγής που έχει να κάνει με την αλλαγή στην, στον αισθημερισμό της εξουσίας μεταξύ της Νέας Ευρώπης που είναι η υποοικοδόμηση και κάθε μιας ε, από τους, καθενός από τους λαούς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ένα νέο κράτος ε, για να γίνουμε καλύτεροι ως Καταλωνία και για να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε στον τομέα των οικονομικών, των πολιτισμικών και των κοινωνικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άκερ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ. Στις 16 Αυγούστου μπήκαν μέσα ε, σε ένα κοντέινερ, λοιπόν και βγήκαν στην εκλογική μου περιφέρεια αφού κρύφτηκαν εκεί δυστυχώς ένας από αυτούς έχασε τη ζωή του. Έχουν από εκείνη τη στιγμή ζητήσει άσυλο και αυτό δεν θα ήταν σωστό να τους δοθεί και θα σας πω γιατί. Ε, εμείς σας δημιουργούμε προηγούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε σημεία εισόδου ε, απαράδεκτα και θα βοηθήσουμε έτσι, θα δώσουμε κίνητρα σε μετανάστες να έρχονται με εμπαρευματοκιβώτια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι πραγματικά αρνητικό και άδικο ε, για τους για τους εκλογείς της περιφέρειάς μου, για τους κατοίκους της περιφέρειάς μου. Ο κύριος έχει το λόγο. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ ενωμένη. Τα κράτη της Ευρώπης πολεμούσαν μεταξύ τους. Αλλά αυτό έχει αλλάξει. Τώρα η Ευρώπη με την κατοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μηδενική οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο λόγος για τον οποίο εμεί δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αντίθετο της Ευρώπης. Το κοινοτικό κεκτημένο είναι το αντίθετο των ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό <clears throat> το οποίο είναι καλό στην Ευρώπη το κάνει κακό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί το πρώτο χαλιφάτο δεν γίνεται στη, στο Ιράκ. Το βλέπουμε στην Νότια Γαλλία. Και πρέπει να το τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεχνητό προϊόν και σταματάει την ανάπτυξη της Ευρώπης. Για όλα αυτά φταίει η Ευρώπη και το κοινοτικό κεκτημένο. Ευχαριστώ κύριε Κόρδιν Μίκε κύριος Μικρό. Μικρό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα ε, σε μια χρονοβόρα διαφωνία, νομική διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ιρλανδικών κατασκευαστικών εταιριών που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με τις πολωνικές αρχές τα τελευταία χρόνια από το 2012 συγκεκριμένα ε, και έχουμε χάσει και 250 εκατομμύρια ευρώ, πολλές θέσεις εργασίες ε, λόγω κακών ε, συνθήκων δημοπράτησης έργων και προκήρυξης διαγωνισμών. Έχουν σταλεί επιστολές και από πέντε άλλες χώρες προς πολιτικές αρχές. Τρία πράγματα θα με ενδιαφέραν. Πρώτα απ' όλα η αρχαιοδοπία της Πολωνίας να αντιμετωπίσει καταγγελίες δίκαια και ειλικρινώς. Δεύτερον, οι πολωνικές αρχές αμέσως θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες διαδικασία ανεξάρτητη ε, διαιτησία για την επίλυση τη νομική αυτή διαφορά. Και τρίτον, στρέφομαι στην Κομισιόν. Έχουμε έναν επίτροπο απόψε. Θα πρέπει, θα πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό πολύ κοντά. Μιλάμε για διαθροτικά ταμεία, για κονδύλια, για λεφτά των φορολογουμένων. Και θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα κονδύλια δαπανώνται, διατίθενται μέσω δημοπράτηση ε, σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέις. Λέω πρόεδρος, επόμενη είναι η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η διαβούλευση για το είδωρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους από το Κοινοβούλιο αυτό πήραν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη του και με τους πόρους του, αλλά όχι όμως με αποκλειστικό γνώμονα το εμπόριο. Στην πόλη μου στο Λονδίνο είδαμε τρομερές αυξήσεις και αυτό ήταν ε, καρπός φυσικά των ιδιωτικοποιήσεων. Η εταιρεία που ελέγχει την διανομή του ύδατος πλήρωσε άνω των 100 εκατομμυρίων μέρισμα στους μετόχους της μόνο για τον προηγούμενο χρόνο. Και υπάρχουν προβληματικές εμπορικές πρακτικές από πλευράς των επιχειρήσεων αυτών και υπάρχει έλλειψη νομικής βάσης για τη δραστηριότητά τους όπως και έλλειψη αποδείξεων ουδετερότητας για τη σωστή τους λειτουργία. Η Βρετανική απάντηση δεν ήταν η σωστή. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα εδαφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε χώρες της Ευρώπης όπως είναι της ε, χώρας των Βάσκων, της Καταλωνίας και της Φλάνδρας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως και αυτό της Σκοτίας. Δεν πρέπει να εμποδίσουμε τους πολίτες να αποφασίσουν και να συζητήσουν. Πρέπει να έχουμε πολιτική δημοκρατία, διάλογο, συμφωνίας και κύρωση από τους πολίτες. Γι' αυτό θέλω να διεκδικήσω το περιεχόμενο της δήλωσης του Στρασβούργου, ώστε τα δικαιώματα όλων των πολιτών θα πρέπει να τυχαίνουν σεβασμού όταν κάποιο κράτος αρνείται να δεχτεί κάτι τέτοιο. Οι εδαφικές εντάσεις είναι αποτέλεσμα της κάμψης των εθνικών κρατών και της θέλησης πολλών από εμά να δημιουργήσουμε την Ομοσπονδιακή Ευρώπη, ένα εγχείρημα για το οποίο εργαζόμαστε εδώ και δεκαετίες. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπιλμπάου Παραντίκα. Κύριος Κάρση. August the 31st last March. 31 Αυγούστου ήταν επέτειος ε, της ε, κατάπασης του πύρους από τον ε, Ήρα. Υπήρξαν βέβαια κάποια προβλήματα τελευταία. Ε, Παρ' όλα αυτά επετεύχθη η, η, Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής όπως γνωρίζουμε πριν πολλά χρόνια και υπήρξε ειρήνευση. Ο ειρηνευτικό διάλογος οδήγησε σε μεγάλη πρόοδο. Τελευταία έχουμε κοινωνικό διάλογο ανεπαρκή δυστυχώ στη χώρα μου και η Ιρλανδική κυβέρνηση, κυρίως η Βρετανική όμως, έχουν αποστασιοποιηθεί από αυτό το διάλογο. Ε, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν υπόψη του, ε, εφόσον στήριξαν, στήριξαν αυτή την ενευτική διαδικασία ότι τα τελευταία συμβάντα με τις παρελάσει ε, στην Ιρλανδία δεν βοηθούν. Ε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές και της Ιρλανδίας αλλά και η Βρετανική κυβέρνηση να συνεχίσει το διάλογο ώστε να εφαρμοστούν πλήρως όλες οι διατάξεις της Συμφωνίας της μεγάλη παρασκευή και όλων των μελλοντικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρθη, να σας υπενθυμίσω ότι ανάβει πάντα ένα λαμπάκι όταν μιλάει ο μιλητής πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να σας διακόψω και να σας ζητήσω να μιλάτε με ανθρώπινη ταχύτητα, μήπως σας καταλάβει και κανένας. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στις τρομερές πλημμύρες οι οποίες ε, πλήττουν την Ινδία, το Πακιστάν και το, το χωρισμένο κράτος του Κασμίρ. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς, έχουμε εκτοπισμένους και φαίνεται ότι θα συνεχίσουν αυτές οι πλημμύρες. Είναι περίπου οι χειρότερες ε, πλημμύρες που έχουν πλήξει το Κασμίρ εδώ και δεκαετίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Κασμίρ είναι μια ε, καυτή περιοχή και είδαμε πολλές, ε, πολλά επεισόδια στη γραμμή ελέγχου μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά θα πρέπει <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι κατά τη διάρκεια των πλημμυρών θα δοθεί υποστήριξη και από τις δύο κυβερνήσεις της Ινδίας και του Πακιστάν και θέλω να ζητήσω η Ευρωπαϊκή Ένωση να, ζητήσει, να βοηθήσει την προσέγγιση των δύο αυτών χωρών για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την πολιτική προστασία. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά αυτές οι δύο κυβερνήσεις και να εργαστούν προς το καλό των ε, λαών τους και όχι να συνεχίζεται αυτή η άσκοπη σύγκρουση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Η οικονομική κρίση στην Ιταλία σε σχέση με την κρίση της μετανάστευσης θα δημιουργήσει προβλήματα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν οικονομικά προβλήματα και που δεν καλύπτονται τα δικαιώματά τους. Η απελπισία αυτών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κινδυνεύσουν τη ζωή τους τους οδηγεί στο να διασχίζουν την Μεσόγειο μέσα σε ε, παλιές ή ε, μη φουσκωτές βάρκες. Εμείς δίνουμε πάρα πολύ ε, λίγα χρήματα σε ένα σύστημα ελέγχου των μεταναστευτικών ροών το οποίο δεν είναι διαφανές και παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε καλύτερα την διαχείριση των ευρωπαϊκών πιστώσεων στα κράτη-μέλη που στοχεύουν σε αυτό, το, σε αυτό το πεδίο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους έτσι ώστε οι μετανάστες να μπορούν να διασχίσουν την θάλασσα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ευχαριστώ κυρία Φεράρα. Ο κύριος Παπαδάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ οι αποφάσεις της πρόσφατης συνόδου του νατο στην ουαλία στρέφονται ενάντια στους λαούς γιατί εντείνουν την επιθετικότητα της υπεριαλιστικής συμμαχίας αυξάνουν τους κινδύνους γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου που θα πληρώσουν ακριβά οι λαοί με το αίμα τους το αποδεικνύουν ήδη οι στρατιωτικές ασκήσεις νατο ηνωμένων πολιτειών και ευρωπαϊκής ένωσης στο έδαφος της ουκρανίας κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με την καπιταλιστική ρωσία για το μοίρασμα αγορών ενεργειακών πηγών και εδαφών. η σημερινή διάσκεψη στο παρίσι για το συντονισμό της στρατιωτικής δράσης των ευρωνατοικών προθύμων κατά των λεγόμενων τζιχαντιστών που οι ίδιοι εξόπλισαν δίνει όθηση στους σχεδιασμούς για επαναχάραξη των συνόρων και γενίκευση της αντιπαράθεσης στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί στρατηγική επιλογή της ευρωπαϊκής ένωσης η ακόμα μεγαλύτερη διασύνδεση με το νατο. είναι τεράστιες οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης γιατί συμμετέχει σε όλους τους επιθετικούς σχεδιασμούς ευρωπαϊκής ένωσης και νατο. το κομμουνιστικό κόμμα της ελλάδας απαιτεί να σταματήσει άμεσα κάθε συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στις αποστολές της ευρωπαϊκής ένωσης και του νατο και παλεύει για την αποδέσμευση της χώρας και από την ευρωπαϊκή ένωση και από το νατο για λαϊκή εξουσία και κυριαρχία με ίδιο Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Να σας υπενθυμίσω οι περισσότεροι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο θέλουν φυσικά να πούν περισσότερα πράγματα. Ο κανόνας όμως λέει ένα λεπτό σας παρακαλώ να περιορίζεστε σε αυτό το λεπτό μην προσπαθείτε να μιλήσετε τόσο γρήγορα και να διαβάζετε γιατί χάνονται πάρα πολλά. Οι διερμηνείς δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν. Και εγώ μετά από ένα λεπτό, πέντε λεπτά, πέντε δευτερόλεπτα μετά από το ένα λεπτό είμαι υποχρεωμένος να σας ε, διακόψω. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παραμείνετε στο πλαίσιο αυτό κύριος Στέκης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Ούγγροι της Ρουμανίας ομόφωνα είναι υπέρ της αυτονομίας ε, του ΣΕΚΕΙ. Αλλά οι κυβερνήσεις είναι κατά της αυτοδιάθεσης ε, των μειονοτήτων και υπάρχει προπαγάνδα κατά των προσπαθειών για το μισό εκατομμύριο των Ούγκρων ε, από την Τρανσιλβανία που θέλουν ε, αυτονομία. Η, τα ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ρουμανίας ε, χρησιμοποιεί την, τις μεθόδους της κομμουνιστικής αστυνομίας για να πέσουν στο κενό αυτές οι προσπάθειες οι απόλυτα θεμητέ προσπάθειε των Ούγγρων ε, τη Ρουμανία και γι' αυτό ζητούμε του Ούγγρου τη Τρανσυλμανία να του προστατέψετε από τι επιθέσει που δέχονται και να στηρίξετε τι προσπάθειέ του για αυτοδιάθεση. Ευχαριστώ κύριε Τεκέσου. Ο επόμενο ομιλητής, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το απόγευμα συζητήθηκε το κατά πόσο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της Ουγγαρίας στην Ολομέλεια. Είπε ένα συνάδελφος ότι δεν υπήρχε τίποτα το καινούργιο για την κατάσταση αυτή. Ναι, μα υπάρχουν νέα στοιχεία. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτής επέκρινε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι δεν μιλάμε μονάχα για ένα θέμα το οποίο <clears throat> αφορά την Ουγγαρία. Αυτό αφορά όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά ένας Πρωθυπουργό χρησιμοποιεί την εξουσία του και τη δύναμή του για να ε, υποσκάψει τις ε, αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τη χρησιμοποιήσει προς το δικό του συμφέρον. Εμείς ως Ευρωβουλευτές έχουμε την υποχρέωση να ορθώσουμε το ανάστημά μας εναντίον αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίγκερ Μίλλερ. Πολύ καλό ήταν που τελειώσατε εγκαίρω τον ε, λόγο σας. Ο κύριος Μα... Μαριάς. Μαριάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αγόρασε κατά τη διάρκεια της κρίσης ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στη δευτερηγενή αγορά με έκπτωση τουλάχιστον 40%. Έτσι η ΕΚΤ κατέβαλε 35 δις ευρώ πλην όμως απαιτεί να εξοφληθεί η ονομαστική αξία των ομολόγων αυτών που ανέρχεται σε 53 δις ευρώ δηλαδή κέρδος 22 δισεκατομμύρια ευρώ. με τον τρόπο αυτό ο κύριος ντράγκη και η παρέα του πουλώντας αέρα κοπανιστό κερδοσκοπούν ασύστολα και ανενδίαστα σε βάρος του φτωχοποιημένου ελληνικού λαού. μόνο για φέτος ο ελληνικός λαός θα πληρώσει καπέλο στην ΕΚΤ 4 δισεκατομμύρια ευρώ και για τον λόγο αυτό η μνημονιακή κυβέρνηση στην αθήνα έχει επιβάλει δυσβάστακτους φόρους στην ακίνητη περιουσία των ελλήνων με τον έμφυα. ο ρόλος της ΕΚΤ όμως δεν είναι να κερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης. έτσι είναι και νόμιμο και ηθικό να κουρευτούν τα ομόλογα αυτά της ΕΚΤ και να πληρωθεί από την ελλάδα μόνο το κεφάλαιο που κατέβαλε η ΕΚΤ για να αγοράσει τα εν λόγω ομόλογα συν ένα επιτόκιο 0,15%. Ευχαριστώ κύριε Μαριά. Και τώρα η κυρία Χάρκιν. Κύριε Πρόεδρε, τον ε, Ιούνιο το Συμβούλιο αποφάσισε να σπάσει τον σύνδεσμο ανάμεσα στις τράπεζες και τα δημόσια χρέη. Αυτό δημιούργησε μια νέα κατάσταση στο δημοσιονομικό πεδίο στην Ιρλανδία και επέτρεψε ταυτόχρονα και την ανακεφαλαιοποίηση των Ιρλανδικών τραπεζών. Λίγο μετά όμως, ε, μια κοινή δήλωση της Μέρκελ ε, και κάποιων άλλων είπε ότι η ε, Ιρλανδία είναι μια ειδική περίπτωση και κανονικά θα έπρεπε να υπάρξει μια κάποια περίοδος αναδρομικής στις ρυθμίσεις που είχαν γίνει, αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει τίποτα και η Eurostat επιβεβαίωσε ότι η Ιρλανδία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κάτω του 1% του πληθυσμού, έχει αναλάβει το 43% του κόστους διάσωσης των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να διαψεύσει τις ε, υποσχέσεις της και θα πρέπει να, να ανακεφαλαιοποιηθούν οι, οι Ιρλανδικές τράπεζες διότι αλλιώς οι συνέπειες θα είναι για όλους άσχημες. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Η κυρία Μπόιλεν. ο Άμπραχα Μαχαλάου, πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνελήφθη τον Αύγουστο του 2013 σε σύγκρουση μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Μόρς. Εξακολουθεί να είναι σε μια Αιγυπτιακή φυλακή χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που κατατέθηκαν εναντίον του. Εξακολουθεί να βρίσκεται να κρατείται σε φρικτές συνθήκες μεταξύ των οποίων σωματική κακοποίηση. Οι Amnesty International και άλλοι οργανισμοί έχουν εξ, ακριβώς την κατάσταση του κυρίου Άμπραχαμ και δεν έχουν βρει λόγους για την κάτσή του. Επρόκειτο να ακουστεί σε ένα δικαστήριο η υπόθεσή του μέσα σε αυτές τις μαζικές δίκες που δεν έχουν νομική υποστήριξη κρατούμενη, αλλά λόγω των ε, διαδικασιών αυτών οι δικηγόροι του αποχώρησαν και τον άφησαν στην φυλακή και δεν μπορεί να συνεχίσει την παιδεία του ή να ανακτήσει την ελευθερία του. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει την απελευθέρωσή του και ο νέος ύπατο εκπρόσωπο να εξασφαλίσει, η νέα εκπρόσωπο να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό ότι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι για την υπόθεση. Ευχαριστώ κύριε Μπόιλεν. Τώρα ο Μάρκ. Dámy Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον προπολογισμό, ε, για να συζητήσουμε τον προπολογισμό ε, της ε, Ένωσης, 150 δι αξία. Αυτά τα 150 δι βγαίνουν όμως από τις τσέπε των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Ίσως κάποιοι πιστεύετε ότι αναδιανέμοντας τους πόρους αυτούς από τις Βρυξέλλες βοηθάμε στο να ζήσουν οι πολίτες καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό είναι λάθος όμως. Πιστεύω το αντίθετο ισχύει. Η αναδιανομή των πόρων βλάπτει την οικονομία, αυξάνει τη διαφθορά και το χρέος. Οι επιδοτήσεις είναι χρήμα που δίνεται στις επιχειρήσεις σε βάρος κάποιου άλλου όμως. Η επιχείρηση που παίρνει την επιδότηση είναι αυτή που βγαίνει κερδισμένη. Όσο μεγαλύτερη ανδιανομή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφθορά. Τρίτον, οι πιο φτωχές χώρες, κυρίως αυτές, να χρεώνονται όλο και περισσότερο για να πάρουν χρήματα ώστε να συγχρηματοδοτήσουν αυτές τις επιδοτήσεις. Κατά την άποψή μου η αναδιανομή των πόρων είναι επιζήμια προς την οικονομία και δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαχ. Η κυρία Κλούν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα μικρά περιφερειακά τοπικά αεροδρόμια έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Και θα ήθελα η Κομισιόν να εστιάσει την προσοχή της σε αυτά τα αεροδρόμια και να εξασφαλίσει ότι αυτά τα αεροδρόμια μπορούν να είναι οι λοκομοτίβες των περιοχών τους και να μπορέσουν να ευνοήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών ώστε οι περιοχές αυτές να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική αγορά και να έχουν συναλλαγές εμπορικές με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν όλο και πιο σημαντικό να μπορέσουν να υπάρχουν αυτά τα αεροδρόμια και θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει οικουμενική προσβασιμότητα στα αεροδρόμια αυτά. Ξέρουμε ότι όταν μια επιχείρηση επενδύει σε μια περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόσβαση με αεροπλάνο και η παρουσία αυτή είναι το κλειδί και για τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο μεγαλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δίνει και ευκαιρίε απασχόληση. Θα ήθελε η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξουν επενδύσει σε αεροδρόμια. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοφα. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουν υπάρξει ζημίες άνω των 300 εκατομμυρίων ε, ευρώ λόγω των καταρακτοδών βροχών στη Βουλγαρία. Πάρα πολλοί έχασαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, η οικονομία μας υποφέρει και η γεωργία μας θα πρέπει και αυτή να ενισχυθεί. Δυστυχώς η φύση πολλές φορές καταστρέφει και όχι μόνο στην Ανατολική Ευρώπη βέβαια. Στις αρχές του 2014 όμως εμείς αλλάξαμε τον κανονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη βοήθεια για φυσικές καταστροφές. Και στο τέλος του μήνα θα πρέπει να μας δώσει ένα εγχειρίδιο διαδικασιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να καταστήσει την απορρόφηση των πιστώσεων για τέτοιες περιπτώσεις ευκολότερη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει ένα καλό κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Αγιώτο. Ο κύριος Μπούντα δεν είναι παρόν. Ο κύριος Μπλένκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφέρω το πρόβλημα ε, των δικαιωμάτων των Κροατών στη Σερβία. Οι Κροάτες οι οποίοι είναι μειονότητα είναι 57.000. Ε, ο κύριος Νίκολιτς έκανε μία δήλωση ότι θα πρέπει κυριλικά να... Ε, και το κυριλικό να χρησιμοποιούν και οι Κροάτες στη Σερβία και αυτό αποτελεί βέβαια διακριτική μεταχείριση, δεν είναι καλή πολιτική και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, έλθει σε συνεννόηση στο πλαίσιο του κεφαλαίου 23 και του κεφαλαίου 24 των δεξιακών διαπραγματεύσεων και να θέσει το ζήτημα αυτό στον δρόμο της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ε, ξεκαθαριστεί γιατί θέλουμε να υπάρχουν και κονδύλια για την εκπαίδευση των ε, κρατών στη Σερβία. Να είναι τα χείριδιά τους δηλαδή στη, στο δικό τους, στη Καπούτο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κρίση των απορριμμάτων στο νότο της Ιταλίας είναι κάτι το κυκλικό το σύστημα απορρόφησης δυστυχώς δεν λειτουργεί παρά την καλή βούληση των τοπικών ε, πληθυσμών που ανταποκρίθηκε στα πλαίσια της διαφοροποιημένης περισυλλογής των αποβλήτων. Θα πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο αυτό γιατί έτσι και αλλιώ έχει παραπεμφθεί η Ιταλία για τα θέματα των επικινδύνων αποβλήτων. Ε, υπάρχουν πάνω των 400 παρανόμων χωματερών και πάρα πολλά άλλα σημεία εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και απορριμμάτων, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον στο περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να αλλάξει και η παρέμβαση η οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, με την εφαρμογή των κανόνων της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας, κάτι το οποίο ε, περιλαμβάνει την ανάληψη ευθυνών και από πλευράς των παραγωγών των διαφόρων προϊόντων και από πλευράς των καταναλωτών αλλά και των τοπικών αρχών. Αυτό θα σώσει από ένα δράμα τις τοπικές κοινότητες. Ευχαριστώ. Άλλους δύο έχω. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Σλοβενία έχει καταφερθεί κατά της έλλειψης ε, διαφάνειας σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στον κόλπο της στεριές της. Πάνω από 100.000 άτομα ζουν σε αυτή την περιοχή. Είναι δύο σημαντικά τα λιμάνια εκεί, το Κότορ και Κόπορ και η Τριέστη. Και είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τουρισμό αυτή η περιοχή. Το να υπάρχουν σταθμοί με ενέργειες με φυσικό αέριο πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο ιδίως η διαδικασία. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Σλοβενίας δεν συμπελήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό εμείς περιμένουμε από την Ιταλία, την Σλοβενία και την Κροατία να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για την ε, τοποθεσία αυτών των σταθμών ενέργειας που πρέπει να τηρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Μπόγκοβιτς. Και τέλος, ο κύριος Πρέδα για να κλείσει τη διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να διαβάσω μία δήλωση του Πρωθυπουργού. Μετά από δέκα χρόνια καθεστώτος Μπασέσκου ε, έχουμε καταστάσεις οι οποίες μοιάζουν με τις επιπτώσεις ε, της ναζιστικής κατοχής ε, στην χώρα. Οι σοσιαλιστές συνάδελφοι συμφωνούν με αυτά τα οποία λέγονται. Μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα τέτοιο καθεστώς. Υπάρχει η περίπτωση να δεχτούμε τέτοιου είδους κριτικές απέναντι σε μια κυβέρνηση, είτε προέρχεται από σοσιαλιστές είτε από συντηρητικούς, να συγκρίνεται με τους ναζί, τους κυβερνήτες της χώρας σας, τους δημοκρατικά εκπλεγμένους. Αν η απάντησή σας είναι όχι, τότε να το πείτε ξεκάθαρα, γιατί ο Πόντα, ο Πρωθυπουργό θέλει να γίνει πρόεδρος της χώρας και δεν μπορούμε παρά να τον εμποδίσουμε. Οι πολίτες της Ρωμανίας δεν θα το επιτρέψουν αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ούτως έχει τελειώσει η διαδικασία ομιλιών ενός λεπτού βαστού του άρθρου 163. Η επόμενη συνεδρίασή μας λαμβάνει χώρα αύριο από τις 9 ως τις 2 ε, και από τις 3 έως ε, τις 8.30. Ε, Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος της συνεδρίασης.